Uh, Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα για συζήτηση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρούνται δεκτά. Είναι διαθέσιμη η διευμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός από γοηδελικά και ε, τη γλώσσα της Μάλτας. Τώρα μέσω της γραπτής διαδικασίας της 5 Οκτωβρίου οι συντονιστές συμφώνησαν να συζητήσουν τη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ για την εφαρμογή των συνθήκων σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία 18-2022. οι συντονιστές συμφώνησαν με την επιστολή η οποία απεστάλλει γύρω από τις αρμοδιότητες σχετικά με την απαγόρευση της διάδοσης υλικού τρομοκρατικής συνάφειας ε, στο διαδίκτυο. Τώρα για τους εισηγητές, ο κύριος Κλοντ Μοράζ είναι εισηγητής για τους ε, διαμεσοφιλικούς, για την έκθεση για τους, για τους διαμεσοφιλικούς πολίτες. Λοιπόν, συμφωνούν οι συνάδελφοι με τις συστάσεις των συντονιστών γενικότερα. σχετικά με την τροπολόγηση του, της ε, πρότασης του 2016 κάθετος 1965 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με την προσθήκη του Πακινστάν στον πρώτο κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνεται στην προσθήκη. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2018 το Συμβούλιο εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του και τον Οκτώβριο του 2018 έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση για την υιοθέτηση του προγράμματος εργασίας για το 2018. η παραλαβή των συγκεκριμένων προτάσεων έγινε στις 18 του μηνός και οι αντιρρήσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 23. 10 παρα 20 να θυμίσω στους συναδέλφους ότι θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας τις κάρτες σας. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις σε σχέση με τα πρακτικά θεωρούνται επίσης δεκτά. Έχουμε τώρα την συνάντηση με την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Να καλωσορίσω την κυρία Φεράρα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στα πλαίσια της συνεργασίας με το άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 45. Έχετε το λόγο, κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ευχηθώ σε όλους μια καλή συνεργασία πάνω σε μια τόσο σημαντική έκθεση. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βάιντεν Χόλτσα και την κυρία Χάουταλα. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτζερ έχει το λόγο. Έχουμε ένα εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας οι δύο εισηγητές, πρόεδρες, συνάδελφοι από τις δύο επιτροπές στα πλαίσια του προγράμματος για τη δικαιοσύνη προωθούμε τα δικαιώματα των πολιτών στον τομέα ακριβώς των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, στα πλαίσια του χώρου δικαιοσύνης, κάτι το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο κράτος δικαίου, ιδιαίτερα για τις διασυνοριακές δράσεις. Έχει τρεις βασικούς στόχους το πρόγραμμα. Πρώτον, στον τομέα των ποινικών το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει και διευκολύνει την δικαστική συνεργασία, προωθεί το κράτος δικαίου, λαμβάνει υπόψη το ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή ε, ε, βοήθεια προς τα κράτη για την κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με τέτοια θέματα και τρίτον ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης ε, ε, και προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων. Απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ε, μέσω της επένδυσης σε, στις επαγγελματικές κατηγορίες που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρόγραμμα Justice λοιπόν θέλει ε, νομίζω όμως κάποιες παρεμβάσεις για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλύπτονται από τις προβλέψεις του. Ε, περιλαμβάνονται επίσης και χώρες τρίτες όπως οι χώρες ΕΖΕΣ, χώρες της γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να είναι αποτελεσματικά εφάκτο λειτουργικό και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία ε, θα έλεγα σε επίπεδο διασυνοριακό ε, πρέπει να καταστούν λειτουργικότερα. Υπάρχει το πρόγραμμα Rights and Values, αξίες και δικαιώματα. Ε, ιδιαίτερα στον τομέα των δικαιωμάτων και του προγράμματος Europe for Citizens. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανάμεσα στα προτινόμενα προγράμματα και κάποιες ε, Σκοτεινέ θα έλεγα περιοχές. Η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων είναι κάτι επίσης το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. αν δεν κάνω λάθος, ε, η εισηγήτρια προτείνει την αύξηση ε, των πιστώσεων. Αυτό είναι σωστό προφανώς, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς οι ανάγκες στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να καλυφθούν. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την τεχνική δομή των προτάσεων. Καλό θα ήταν να δούμε αν οι προσθήκες στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι τμήμα των συνολικών προτάσεων. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος ένα κομμάτι βασικό της έκθεσης να είναι απλό παράρτημά της. Θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο θέμα της εμπορίας ε, όλα αυτά απαιτούν ε, ειδικέ γνώσεις και ειδικέ ικανότητες, οπότε θα πρέπει να καταστήσουμε τις αρχές ικανές να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η σωματεμπορία είναι μια ποινικά κολάσιμη δραστηριότητα φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες και η αντιμετώπιση της απαιτεί περισσότερους πόρους. Απαιτείται επίσης περισσότερη διαφάνεια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε την διαφάνεια έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι καλύπτονται από το πρόγραμμα να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Η ε, χρηματοδότηση της διευκόλυνσης προσφυγής στη δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι κάτι το αντικειμενικό που να αρμόζει στους κανόνες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Τα θύματα θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες και να έχουν με καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αν και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αρμοδιότητα στα πλαίσια μιας εθνικής δικαιοδοσίας για διασυνοριακές υποθέσεις, τα δικαιώματα των θυμάτων δεν καλύπτονται απόλυτα σωστά. Θα πρέπει λοιπόν τα θύματα των διασυνοριακών ε, εγκλημάτων ή ποινικών, ε, ποινικά κολάσιμων πράξεων να είναι δυνατόν να διώκονται ε, και νομίζω ότι όλα αυτά που είπα είναι κάποια παραδείγματα στα οποία θα πρέπει να σταθούμε θα ήθελα να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο ε, το αν θα πρέπει να τροπολογήσουμε τις προτάσεις αυτές ε, περαιτέρω σε συνεργασία με τον κύριο Βάιντεν Χόλτζα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα, ο κύριος Βάιντεν Χόλτζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό γιατί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ε, στους πολίτες πρέπει να είναι βασικό στόχος για μας. Πρέπει να εμπιστεύονται τα νομικά μας συστήματα. 200 ευρώ έχει, 200 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα δικαιοσύνη. Σε αυτό καταλήξαμε έπειτα από αξιολογήσει που είχαμε και έπειτα και από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους. Πώς ε, τα οικοδομήσαμε τα προγράμματα. Έγινε μια εσωτερική εξολόγηση των ε, τρεχών των προγραμμάτων, από την οποία προέκυψε ότι οι στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν και ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την ε, επιδίωξη να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Επίση, σημαντικό στοιχείο είναι η ενωσιακή προστιθέμενη αξία στην ενδιάμεση αξιολόγηση και χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση των ε, ετούντων, απλούστευση των κανόνων και όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα συμπεριλάβουμε στι νέε μα προτάσει. Επίση, έγινε και μια δημόσια διαβούλευση η οποία υποστήριξε πραγματικά την επιλογή της Κομισιόν να επικεντρωθούμε στις αξίες, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στο γεγονός ότι η δημοκρατική συμμετοχή, το κράτος δικαίου, γενικά οι ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να ενισχυθούν και να τονιστούν. Επίσης, υπάρχει προστιθόμενη αξία του προγράμματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δικαιώματα και οι αξίες και τα δικαιοσύνη επιτυχάνουν ακριβώς αυτό. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η δικαστική συνεργασία. Χρειάζονται περισσότερες συμπράξεις μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και αυτό είναι επίσης ένας από τους στόχους της Κομισιόν. Τώρα για το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Αυτό που προκύπτει και από τη μελέτη επιπτώσεων είναι πρώτον ότι χρειαζόμαστε συνέχεια με το τρέχον πρόγραμμα γιατί οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη. Επομένως η, Κομισιόν, η πρόταση της Κομισιόν αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό, στο να εξασφαλιστεί η συνέχεια των ε, τρεχουσών δραστηριοτήτων, η συνέχιση τους δηλαδή, να υποστηριχθεί η δικαστική συνεργασία σε ποινικά και αστικά ζητήματα, να προωθηθεί το κράτος ε, δικαίου, να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η κατάρτιση και η εκπαίδευση δικαστών, προκειμένου να ε, ενισχυθεί και η γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα ένδικα μέσα εν γέννη, να, βελτιωθούν η, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και να προστατευθούν τα δικαιώματα των θυμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα, ε, οι βασικότεροι στόχοι του προγράμματος. Τι δραστηριότητε θα χρηματοδοτούνται. Έχουμε ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, αμοιβαία μάθηση, μέσω ανταλλαγής, των πρακτικών, αναπτύσσουμε ε, πληροφορία Ότητα της νομολογίας και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το διαχωρισμό εξουσιών σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτή δεν ήταν καθόλου ιδέα ε, της ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώρισης. Ακριβώς αντίθετα, η ιδέα ήταν να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη. Και αυτό τι σημαίνει, ότι οι δικαστές θεωρούν δεδομένο ότι σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μια, ένας βασικός σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων Υπάρχει εξαρτησία της δικαιοσύνης και υπάρχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα για να διορθωθούν προβληματικές αποφάσεις ενός δικαστηρίου στην ίδια χώρα. Στο βαθμό που ο δικαστής ο, του κράτους μέλους, το οποίο εμπλέκεται σε μία υπόθεση δικαστικής συνεργασίας, αξιολογεί την ε, σημασία, την, ε, την, την ποιότητα των αποφάσεων του άλλου κράτους, των δικαστηρίων του άλλου κράτους μέλους, στην πραγματικότητα αρνείται την, τον ίδιο το χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος λοιπόν της συνεργασίας θα πρέπει να τονιστεί και στο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη και στη δικαστική κατάρτιση και εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο, α όχι, ο κύριος κρυπακ Για δύο λεπτά. Και εγώ εκπροσωπώ το σκιώδη εισηγητή μας. Λαμβάνουμε υπόψη τα κίνητρα της πρότασης της Κομισιόν. Ο κύριος Μανταγκούρεκ έχει αντίστοιχες ανησυχίες για τη δημιουργία του νέου προγράμματος δικαιοσύνης, όπως είχε για τα δικαιώματα και την... ή μάλλον για το πρόγραμμα ε, δικαιωμάτων και αξίας όπου η δουλειά της ΛΥΠΕ έχει προχωρήσει. Η κυρία Βαλέρο έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς της Επιτροπής ΛΥΠΕ για το θέμα αυτό. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο, λέμε, τους περισσότερο, περισσότερο ΜΚΟ ε, που προωθούν τις ευρωπαϊκές προσθέμενες αξίες σε αυτό το συρρυκνούμενο χώρο ε, ελευθερίας και δικαιοσύνη σε κάποια κρατημέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι μια απόπειρα να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια ε, ω ήπια δύναμη εναντίον κάποιων χωρών, λέει ο σκιώδη εισηγητή, και μπορεί να δημιουργήσει διαιρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η κανονιστική φύση των αξιών του άρθρου 2 τη συνθήκη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείει και το τονίζω το να ερμηνεύουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις ε, όπως θέλουν τις διατάξεις. Επίσης, συχνά, η πρόταση της ε, Κομισιόν για, την, ε, για το πρόγραμμα δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο δεν θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιηθούν ε, εναντίον των απόψεων ορισμένων ομάδων σε κάποια κράτη-μέλη. Μιλάμε για κοινού δημοσιονομικού πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει, η συμπρόεδρο μας θα κάνει και αυτή μια παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές φορές ε, Έχουμε παραπονεθεί για την έλλειψη εμπιστοσύνη ε, στα κράτη-μέλη στον τομέα της δικαστικής ε, συνεργασίας. Ε, και αυτό περιορίζει τις δράσεις για την καταπολέμηση της δημοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ακόμα μια φορά ότι η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική στον τομέα αυτό. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη αμοιβαία αναγνώρισης. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη κάθε φορά που μιλάμε για εργαλεία συνεργασία συγκεκριμένα. για να υπάρχει πραγματική εφαρμογή αυτής της αρχής, της αμοιβαίας αναγνώρισης δηλαδή, ακόμα και στη φάση της διαπραγμάτευσης των μέσων αυτών, θα πρέπει να διευκολύνουμε την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κανονιστικών πράξεων, ε, ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που μπορούν να μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να της κάνω εξή ερώτηση. Μπορείτε να μας Δώστε περισσότερες λεπτομέρειες ποιες δράσεις σκοπεύετε να προωθήσετε ούτω ώστε να εγγυηθείτε αυτή την εμπιστοσύνη και την αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Κατανοούμε ότι υπάρχει κοινός χώρος εργασίας για διάφορα τμήματα του προγράμματος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας και θέλουμε να συνεργαστούμε ως προς αυτό με το Κοινοβούλιο. Όπως είπα, το πρόγραμμα βασίζεται σε μια αναλυτική παρουσίαση, βασίζεται επίσης σε μια μελέτη των επιπτώσεων της πιθανής εφαρμογής του και νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από το σεβασμό των αξιών που απαιτούμε. Μιλήσαμε Πάντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 31. Ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε πια. Εγκρίνεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 75. Ψηφίζουμε. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίπτεται. 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές 35. Η... Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 για την εντολική σκέψη 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Αιτιολογική σκέψη 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Για την αιτιολογική σκέψη 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ.